Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, να αρχίσουμε τη συνεδρίασή μας σήμερα. Πρέπει να σας ε, ρωτήσω αν έχετε να προτείνετε κάποια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη για σήμερα. Όχι. Καλώς. Δεν έχω και ανακοινώσεις. Ούτε ανακοινώσεις του Πρόεδρου έχω. Και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει όσον αφορά τα πρακτικά των συνεδριάσεων τη 26η Ιανουαρίου, Δευτέρα Φεβρουαρίου και 9η Φεβρουαρίου, τότε θεωρούνται εγκεκριμένα. Θέλω να υποδεχτώ εδώ τον ε, Ομερπάντο Κιπίκο, που είναι πρόεδρος του Κοινοβουλίου από την Βουλή των Αντιπροσώπων στη Ζάνζιμπαρ στην Τανζανία. Όπως ξέρετε η Τανζανία είναι μια χώρα προτεραιότητα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η το σώμα μας παρακολούθησε τις εκλογές, είναι από τους έξι εταίρους κατά προτεραιότητα για την ανάπτυξη της δημοκρατίας και σχετικών δραστηριοτήτων το 2015. Η σημερινή επίσκεψη είναι το πρώτο βήμα για την ανάπτυξη αυτής της εταιρική σχέσης παρετέρω και προκειμένου να έχουμε και διάφορες πρωτοβουλίες παρακολούθησης. Φιλοξενούμε λοιπόν και την συνέλευση της Ένωσης και τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Είναι μια σημαντική χρονιά για την Τανζανία. Τον Οκτώβριο θα έχει εκλογές. Επίσης προτάθηκε πρόσφατα αλλά αναβλήθηκε ένα δημοψήφισμα. Φαντάζομαι ότι θα μας ενημερώσει ο μας περισσότερο από αυτού. Σήμερα έχουμε μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ακούσουμε τον κύριο Παντούα Μεκυπίκο και να έχουμε ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά τις προετοιμασίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν Ζάνζιβάρ και η Τανζανία εν ώψη των εκλογών εκεί. Αυτή ήταν η σύντομη εισαγωγή μου. Τώρα, αξιότιμε πρόεδρε του Κοινοβουλίου, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, ή κάνω λάθος. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ για να μοιραστώ μαζί σας ε, με την αντιπροσωπεία εδώ της Βουλής των Αντιπροσώπων της Ζανζιβάρης στην Τανζανία και συνοδεύομαι από άλλα πέντε μέλη, συμπεριλαμβανομένου μου και πέντε εξωματούχου. τέσσερις εξωματούχους, συγγνώμη, ένας από του οποίου είναι επικεφαλή τη βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Γιαγιαβή Σαμάτ, και οι λοιποί εξωματούχοι είναι βοηθοί του πρώην ε, Υπουργού τη Ζανζιβάρης, ε, Υπουργού Δικαιοσύνη που κάθεται εδώ Ενδεχομένω μπορεί να σηκωθεί για να τον δούμε ο κύριος Γιαχώδα, παρακαλώ Uh, Τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας είναι ο κύριος Αμπτάλα Γιούμα. Μπορείτε να σηκωθείτε παρακαλώ. Ο κύριος Χαμάτ παρακαλώ. Η κυρία Ουαν Χαφινταμέρ. Η κυρία Ζάρα Αλχαμάτ. Ο κύριος Γιάννη Χαμισαμάτ. Και εγώ που ήδη ο κεφίκιο ε, από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, υπήρξα ε, ομιλητής της ε, Βουλής εδώ και πολλά χρόνια και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικά ζητήματα σε σχέση με την εμπειρία μας από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που έχουμε στη Ζανζιβάρη. Οπότε, επιτρέψτε μου μερικά λεπτά κύριε Πρόεδρε για αυτή την παρουσίαση. Θα ξεκινήσω με ένα μικρό ιστορικό για το σχηματισμό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Ζανζιβάρη. Η κυβέρνηση αυτή Εθνικής Ενότητας προήλθε από τις ε, μη αναμενόμενες ελεύθερες συνομιλίες που οδήγησαν συζητήσεις μεταξύ από τον πρόεδρο της Ζανζιβάρης ε, Πιντούση και τον κύριο Αμάν Αμπτέτ Καρούμι. Ο Γενικός Γραμματέας ε, της τότε αντιπολίτευσης ε, της, ε, του Ενωμένου ε, Μετοπολιτών, ο κ. Σαρίφ Χαμάντ, ο οποίος τώρα είναι πρώτος αντιπρόεδρος της Ανζιβάρη. από τις 15 Νοεμβρίου του 2009. Οι συνομιλίες μεταξύ αυτών Ε, ήταν απόρριτες και κανείς δεν ενημερώθηκε πλήρως. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα μας εξήγησαν αργότερα, ε, αντιληφθήκαμε ότι οι συζητήσεις τους ε, εστιάστηκαν στο ζήτημα ύπαρξης μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας Ε, έτσι ξεκίνησαν οι συζητήσει μεταξύ των δύο πολιτικών κομμάτων, του CCM, το CCM που ήταν το τότε κυβερνών κόμμα και που συνεχίζει να είναι το κυβερνών κόμμα τόσο στην, Τανζανία, στην υπηρετική Τανζανία και στην ε, Ζανζιβάρη και του CUF το οποίο ουσιαστικά συμφώνησε για το σχηματισμό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας. Αυτό συνέβη μετά από διάφορες συζητήσεις και διάλογο μεταξύ των δύο κομμάτων. Ε, συναντήσεις έγιναν σε διάφορους χώρους ε, όπως το Νταρασαλάμ και στον Παλαμόδιο. Εκεί λοιπόν ε, τονίστηκε ότι είναι σημαντικό η Ζανζιβάρη να έχει κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Αυτό είναι σημαντικό διότι Για πολλά χρόνια είχε υπάρξει ιστορικό πολιτικό διέξοδο το οποίο υπονόμευε την ανάπτυξη της Ζεβάρη. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να περάσουμε σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας ώστε να τερματιστεί αυτή η πολιτική αντιπαράθεση και να προωθηθεί η ανάπτυξη της χώρας. Με μια φιλική στάση μεταξύ των δύο βασικών πολιτικών κομμάτων του CCM και του CUF. Μετά από αυτή τη συζήτηση, το διάλογο των δύο επικεφαλής των πολιτικών κομμάτων του Ζανζιβάρη, του πρώην Πρόεδρου της Ζανζιβάρης, του κυρίου Καρούμε και του Γενικού Γραμματέα, του κυρίου Σεριφαμάντ, όπως ήταν ε, ε, Μάλιμ σημαίνει δάσκαλος από τα αραβικά. Συμφώνησαν λοιπόν και μετά έγινε μια πρόταση ψηφίσματος στο Βουλή των Αντιπροσώπων για το πώς θα ε, δημιουργείται μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Έγινε ανταλλαγή ιδεών και η πρόταση για την κυβέρνηση εθνικής ενότητας ε, είχε ως εξής το να υπάρχει μια κυβέρνηση όπου αυτά τα δύο πολιτικά κόμματα από κοινού θα κυβερνούν. Ούτως και πράξαμε. Και έτσι τερματίστηκαν όλα τα προβλήματα που είχαμε. Είναι μια νέα μορφή κυβέρνησης στην Τανζανία. Εδώ στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έχετε ε, κυβερνήσεις και αντιπολίτευση. κυβερνήσει συνασπισμού και ε, αντιπολίτευση, αλλά εμείς επίσημα δεν έχουμε ε, αντιπολίτευση. Θα μπορούσε να αναρριτηθεί κανείς αν η δημοκρατία πολλών κομμάτων είναι τόσο σωστή όσο στη δική μας κυβέρνηση που εμείς δεν έχουμε αντιπολίτευση. Μπορώ να σας πω ότι τα πράγματα λειτουργούν πολύ καλά σε μας. Και είναι σαν να έχουμε αντιπολίτευση γιατί όλα τα μέλη όλων των κομμάτων ε, του κυρίου κόμματο του CCM και του ε, μικρότερου κόμματο του UF, όλα τα μέλη συνεργάζονται μαζί και υπάρχει κατά κάποιο τρόπο μια αντιπολίτευση για όλα τα ζητήματα. Και στα μπροστινά έδρανα ε, όπου κάθονται συνθουσοί υπουργοί ε, Εκεί έκαναν οι υπουργοί του κυρίου κόμματο. Έτσι λοιπόν αυτή η κυβέρνηση συνασπισμού λειτουργεί. Τίποτα δεν υπονομεύει την ύπαρξη πολλών κομμάτων στη δημοκρατία της ε, Ζανζιβάρης και στην Τανζανία γενικότερα. Αλλά αυτή η μορφή κυβέρνησης λειτουργεί μόνο για τη Ζανζιβάρη και όχι για ολόκληρη τη χώρα. Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς ε, γιατί δεν έγινε αυτό για ολόκληρη την Τανζανία, τόσο για την κυβέρνηση της Ζανζιβάρης όσο και για την ε, κυβέρνηση όλης της χώρας. Διότι το ιστορικό υποβάθρο είναι διαφορετικό. Το ιστορικό υποβάθρο που έχουμε στη Ζανζιβάρη μετά από κάθε ε, εκλογική αναμέτρηση η διαφορά ήταν πολύ μικρή. συγγνώμη, η αντιπολίτευση ήταν πολύ μικρή. Οπότε δεν ήταν δυνατόν να λειτουργήσει μια κυβέρνηση με τον αριθμό εδρών. Να σας δώσω το παράδειγμα των εκλογών του 1995, το κυβερνών κόμμα είχε 26 έδρες από τις 50. Οπότε βλέπετε ήταν ε, πολύ ε, στενή αναμέτρηση. Έτσι λοιπόν ε, ήταν σαν μια διελκυστίνδα. Ήταν δύσκολο να λειτουργήσει η κυβέρνηση χωρίς να υπονομεύονται τα αναπτυξιακά έργα που κάνουμε στην Τανζανία. Αλλά ιστορικά το CCM ανέκαθεν νικούσε ε, την πλειοψηφία των εδρών ε, και ε, στην κυβέρνηση της Τανζανίας ε, το κόμμα το οποίο νικάει είναι αυτό που σχηματίζει μόνο του την κυβέρνηση. Τα κερδίζει όλα δηλαδή. Έτσι έχουμε οργανώσει την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Υπάρχουν διάφορες πτυχές. Φυσικά ναι, καθεν είχαν τα πολιτικά κόμματα συζήτηση. Αλλά ε, ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει και δυνατότητα δημοψηφίσματος. Αυτό δεν το κάναμε παλιά απευθείας, διότι το Σύνταγμα μας δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο. Χρειάστηκε λοιπόν να προβούμε σε κάποιες αλλαγές, σε τροποποιήσεις του συντάγματος, ώστε να μπορέσει να δημιουργηθεί η κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Έτσι δίνουμε και στην εκλογική επιτροπή της Ζανζιβάρης την εξουσία να μπορέσει να διαχειριστεί το δημοψήφισμα. Διότι δεν αποφασίσαμε απλά να έχουμε μία ε, κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ε, το περάσαμε από δημοψήφισμα. Για να ολοκληρώσω την παρουσίασή μου, ε, κύριε Αντιπρόεδρε, μπορώ να πω ότι τελικά η διαδικασία που οδήγησε στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας βασίστηκε σε τρεις ε, πτυχές. Έγινε διάλογος και συζήτηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων που οδήγησε στην κυβέρνηση αυτή Εθνικής Ενότητας. Δεύτερον, η πρόταση ψηφίσματο ε, για την κυβέρνηση εθνική ενότητα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Και τρίτον, η τροποποίηση του συντάγματος, που είναι η δέκατη τροποποίηση, που εγκαθίδρυσε την κυβέρνηση εθνική ενότητα. Αλλά και το άλλο που έγινε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό τη δική μου ε, ηγεσία ως ομιλητή, ήταν το να γίνει ένα δημοψήφισμα ως πρόεδρο του Κοινοβουλίου ώστε να γίνει ένα δημοψήφισμα ώστε να δημιουργηθεί η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος που έγινε όπως ε, γίνονται και οι γενικές εκλογές ήταν 66,4% υπέρ της κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 33, κάτι κατά έτσι τροποποιήσαμε το Σύνταγμα λόγω του αποτελέσματος ε, του δημοψηφίσματος που ήταν υπέρ της κυβέρνησης της Εθνικής Ενότητας. Επ' αυτού θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ακούσατε την παρουσίασή μου κύριε Αντιπρόεδρο. Ευχαριστούμε πολύ. Πριν δώσω το λόγο στους συναδέρφους, μήπως θέλουν να ρωτήσουν κάτι, θα ήθελα εγώ να σας ρωτήσω πώς έχει η κατάσταση που ξέρουμε ότι είναι ασταθής στο κέντρο της Αφρικής, στους γειτονές σας και πώς επηρεάζει αυτή η κατάσταση την πολιτική ζωή της χώρας σας. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια για αυτό παρακαλώ. Ο κύριος Η κατάσταση στις γείτονες χώρες στην Ανατολική Αφρική, Κένια, Ουγκάντα, Μπουρούντι, Ρουάντα και Σομαλία που γειτονεύει με την Κένια. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Στα σύνορα Κένια, Σομαλία. Γιατί υπάρχει η al Όλοι τη γνωρίζετε και όλοι ξέρετε τι κάνει στη Σομαλία. Δεν υπάρχει σταθερή κυβέρνηση σήμερα στη Σομαλία. Από πλευρά της Κένια επίσης υπάρχει πρόβλημα με την Al Shabaab, οι οποίοι προκαλούν αστάθεια και ανασφάλεια στη χώρα έχουν συμβεί, τα ξέρετε, πριν από λίγο καιρό διάφορα. 67 έχασαν τη ζωή τους και πρόσφατα 141 έχασαν τη ζωή τους σε μία από τις επιθέσεις. Αυτή είναι η κατάσταση όσον αφορά την Ασαμπά. Στις υπόλοιπες περιοχές πάμε καλά. Γιατί δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. Δεν έχουμε όπως τη Σομαλία που σας είπα. Η Σομαλία είναι μεμονωμένη περίπτωση από την πλευρά της Κένια και μετά. Αυτό που μπορώ κάπως σύντομα να σας πω είναι ότι στην Τανζανία πολιτικά προχωράμε πολύ καλά και ελπίζουμε να έχουμε εκλογέ τον Οκτώβριο που μας έρχεται και δημοψήφισμα τον Ιούλιο φέτος κατά πάσα πιθανότητα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Τάνοκ. Και μετά κύριε Φωτίγα, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να καλωσορίσω ιδιαίτερα την αντιπροσωπεία της ε, Ζανζιβάρης. Πρόκειται για ένα αρχιπέλαγο με το οποίο εμείς ε, το Ηνωμένο Βασίλειο είχαμε μία σημαντική ιστορική σχέση και τώρα φυσικά ως τμήμα της Τανζανίας η νησιωτική αυτή επαρχία εξακολουθεί να έχει ένα σημαντικό ρόλο. Θα ήθελα να αναφερθώ στη ριζοσπαστικοποίηση και τις επιθέσεις που έχουν γίνει από το Βάμσο ιδίως σε εκκλησίες, στην Αγγλικανική Καθεδρική Εκκλησία, σε εστιατόρια και μπαρ. Σε ποιο βαθμό λοιπόν υπάρχει ασφάλεια στα νησιά της Ζανζιβάρης και κατά πόσο αυτή η ανασφάλεια υπονομεύει τον τουρισμό, σε ποιο βαθμό οι νέοι σας γίνονται τζιχαριστές ή πηγαίνουν στη Συρία και το Ιράκ. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ γιατί είναι τμήμα της παγκόσμια, του παγκοσμίου στερεώματος ασφάλειας αυτό το οποίο συμβαίνει στην περιοχή. Ευχαριστώ για το ερώτημά σας. Η ΟΑΜΣΟ είναι ένας φορέας ο οποίος έχει <clears throat> ιδρυθεί ως μια ένωση ατόμων που είναι μουσουλμάνοι βέβαια αλλά δεν έχουν καμία σχέση με το Ισλαμικό κράτος ή οποιοδήποτε παρακλάδι της Αλκάιντα ή της Al-Shabaab. Είναι μια οργάνωση λοιπόν η οποία έχει προέλθει από τη Ζανζιβάρη Δεν θέλαμε να συμβεί κάτι τέτοιο στα νησιά μας. Και η κυβέρνηση της Ζανζιβάρης φυσικά είναι εναντίον της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με τη δράση της Γουάμσο. Αυτοί οι οποίοι λοιπόν έχουν συμμετάσχει στο κίνημα αυτό στο παρελθόν. Βρίσκονται στην, στο, ενώπιον του δικαστηρίου και η δίκη είναι εν εξελίξη. Περιμένουμε λοιπόν το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας. <clears throat> Αλλά μπορώ να πω ότι η Ουάνσο δεν είναι μια ομάδα η οποία συνδέεται με κάποιο πολιτικό κόμμα εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχει σχέση με κάποιο άλλο διεθνή φορέα ή κίνημα ή οργάνωση. Είναι μια ομάδα ατόμων που προέρχονται από τη Ζανζιβάρη και οι δικοί τους ισχυρισμοί ήταν ότι δημιουργηθήκανε γιατί δεν υπήρχε ελευθερία, δεν υπήρχε δίκαιος τρόπος να αντιμετωπιστεί το θέμα των μουσουλμάνων στη Ζανζιβάρη. <clears throat> Μέχρι τώρα όμως η κυβέρνησή μας έχει κάνει προσπάθειες να σταματήσει κινήσεις αυτού του είδους. Και όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν συμμετάσχει σε αυτό το κίνημα είναι στην ενώπιον της δικαιοσύνης και περιμένουμε την απόφαση της δικαιοσύνης. Ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. χρησιμοποιεί μη, μη ευρωπαϊκή κοινοτική γλώσσα. Ο κύριος Κούκαν μάλλον τα λέει στα Σουαχίλη. Μόλις χαιρέτησα τον φίλο μας από τη Ζανζιβάρη. Κάπως δεν τα καταφέρνουν οι διερμήνες από τα Σουαχίλη από ό,τι διαπιστώσαμε. Αλλά νομίζω ότι με κατάλαβε ο... Με κατάλαβε η αντιπροσωπεία της Ζαζιβάρης. Σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω θερμά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την αντιπροσωπεία σας από αυτή την τόσο όμορφη χώρα της Αφρικής. Είπατε ότι θα πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα προσοχή για την δημοκρατία της Τανζανίας. Είναι μια χώρα η οποία δεν εμφανίζεται τόσο πολύ στις ειδήσει. Αυτό είναι βέβαια φιλοφρόνηση προς εσάς γιατί δεν δημιουργείται προβλήματα. Πιστεύω όμως ότι πρέπει να ενισχύσουμε περισσότερο τη συνεργασία μας μαζί σας. Θα λάβουν χώρα μέχρι το τέλος του έτους βουλευτικές εκλογές στην Τανζανία και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποστείλει μια, εκλογική, μια αποστολή εκλογικής παρακολούθησης και αυτό θα είναι μια ευκαιρία να μάθουμε περισσότερα για την χώρα σας και όταν γυρίσει αυτή η αντιπροσωπεία θα είναι πάρα πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία θα μας πούν για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία μας μεταξύ Ευρώπης και της χώρας σας και να αναβαθμίσουμε τις σχέσεις αυτές κατά ένα κλικ. Και συνεχίζει στα σου αχίλια κύριος you very much. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι η Τανζανία συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας έχετε στηρίξει πολύ σε διάφορους τομείς. Όσον αφορά θέματα ανάπτυξης, για παράδειγμα. Επίσης, είναι αλήθεια ότι η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήγε εκεί ο παρατηρητές των εκλογών. Και θυμάμαι ότι το αποτέλεσμα ήταν θετικό. Ελπίζουμε λοιπόν ότι αυτή τη φορά τα εκλογικά σώματα θα προσκαλέσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και πάλι για να έρθουν ως παρατηρητές στις εκλογές και ελπίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Πέρυσι για πρώτη φορά Συνεργαστήκαμε μαζί σας και τώρα υπάρχει θέση στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έρθει παρατηρητή στις εκλογές μας. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή. Ελάτε σας παρακαλώ. Να παρακολουθήσετε τις εκλογές μας. Και ελπίζω ότι θα σας καλέσουν τα εκλογικά σώματα. Παντού. Η κυρία Φωτίγκα τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξοχότατε, εξιότιμοι βουλευτές τη Ζάντζιμπαρ Τανζανία, καλώς ήρθατε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να αναφερθώ λίγο στο ρόλο της Τανζανίας στην περιοχή και γενικότερα στην Αφρικανική Ήπειρο μια που προσφέρει ειρήνη και συμφιλίωση. Θέλω να αφαιρθώ στις συμφωνίες της Αρούσα, αλλά και άλλες προσπάθειες που έχουν γίνει. Εσείς πώς βλέπετε το θέμα της σταθερότητας στην περιοχή, λαμβάνοντας υπόψη τις παραβιάσεις της συνευτικής ε, συμφωνίας συμφιλίωσης της Αρούσα για τον Μπουρούντι εξαιτία των αποφάσεων που πήρε το κυβερνόν κόμμα. Τι δυνατότητα υπάρχει να συνεχίσει η ειρήνη, να υπάρξει μάλλον η ειρήνη μετά από τόσα χώρια, χρόνια εμφυλίου πολέμου σε χώρες όπως είναι το Μπουρούντι, η Ρουάντα και το Κονγκό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση, κυρία μου. Η Τανζανία πάντα ήταν στην πρώτη γραμμή υπέρ της ειρήνης και της ηρεμίας. Τόσο στην Τανζανία την ίδια, όσο και στις γειτονές χώρες. Οπότε αυτά τα οποία έγιναν στο Μπουρούντι και στη Ρουάντα για χρόνια, όντως ήταν μια δύσκολη κατάσταση και για μας. Πρόσφατα Εξαιτίας της τρίτης προσπάθειας ε, για προεδρία στο Μπουρούντι, εμείς στη Δανζανία έχουμε ένα σύστημα δύο πεντετίες στην Προεδρία. Και η κυβέρνηση Τη Τανζανίας. Πιστεύω ότι θα κάνει έκκληση στους ηγέτες των Μπουρούντι να τηρήσουν το Σύνταγμα για δύο θητείες. Νομίζω ότι αυτό λέει τώρα. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα. Γι' αυτό, άνθρωποι. Η Τανζανία ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή υπέρ της ειρήνης και της ηρεμίας. Όχι μόνο μέσα στη δικιά μας τη χώρα την Τανζανία, αλλά και στις γείτονες χώρες. Η Τανζανία πρέπει να θυμηθούμε ότι ήταν στην πρώτη γραμμή και για την ανεξαρτησία. Εμείς λέμε ότι η Τανζανία δεν είναι ανεξάρτητη εάν κάποια άλλη αφρικανική χώρα δεν είναι ανεξάρτητη. Έτσι συνηθίζαμε να λέμε. Γι' αυτό και η Τανζανία είναι πάντα στην πρώτη γραμμή υπέρ της ανεξαρτησίας και της ελευθερίας. Αυτό θέλουμε για όλες τις χώρες. Υπέρ της ειρήνης, της ηρεμίας δημοκρατικά σε αυτές τις διάφορες χώρες που αναφέρατε της Αφρικής. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η κυβέρνησή μας θα δράσει ώστε αυτό το συνεχιζόμενο πρόβλημα στον Μπουρούντι θα σταματήσει. Θα προσπαθήσουμε να συμβουλέψουμε του συναδέρφους μας εκεί για να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Ευχαριστούμε κύριος Μακάλιστερ. Εξοχρωτάτε κυρίες και κύριοι αγαπητοί συναδέλφοι. Χαίρομαστε ιδιαίτερα που βρίσκεστε εδώ μαζί μας. Είμαι Γερμανός και όπως σας γνωρίζετε τα 16 κρατήδια της Γερμανίας έχουν όλα με ε, συμφωνίες συνεργασίας με τη Ζανζιβάρη. Και εγώ θυμάμαι πόσα, σε πόσα έργα προσπαθήσαμε να σας προσφέρουμε αρρωγή και οικονομική βοήθεια. Έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, πότε πιστεύετε ότι θα λάβουν χώρα οι εκλογές. Ή αν δεν το γνωρίζετε, πότε πιστεύετε ότι θα ανακοινωθεί η ακριβή ημερομηνία των εκλογών. Δεύτερη ερώτηση, Πώς θα πηγαίνει η Τανζανία όσον αφορά τον τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ. Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Τανζανίας, κανονικά οι εκλογές ε, λαμβάνουν χώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου κάθε πέντε έτη. Αυτή τη φορά ελπίζουμε λοιπόν να γίνουν οι εκλογές, αν δεν κάνω λάθος, στις 25 Οκτωβρίου φέτος, το 2015. Και ελπίζουμε ότι θα τηρήσουμε αυτή την ημερομηνία, διότι παραδοσιακά τότε λαμβάνουν χώρα οι εκλογές κάθε πέντε χρόνια την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Η τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου λοιπόν αυτή τη φορά θα είναι 25η. Ελπίζουμε λοιπόν να λάβουν χώρα οι εκλογές. Εκείνη την ημερομηνία. Η δεύτερη ερώτηση ήταν, συγγνώμη, ποια είναι τα μελλοντικά σα σχέδια για τον τουρισμό στην όμορφη σας χώρα. Να σας μιλήσω κατά περιοχές και να ξεκινήσω από τη Ζανζιβάρη. έχουμε διαφορετικά οικονομικά ζητήματα στη Ζανζιβάρη και στην υπηρετική Τανζανία. Εμείς στη Ζανζιβάρη για μας ο τουρισμός ε, είναι ο δεύτερος, ε, το δεύτερο υψηλότερο εισοδηματικός παράγοντας ε, μετά από το μετά από το γαρίφαλο. Και έτσι πιστεύω ότι μπορούμε ε, να δικήσουμε τα πράγματα αρκετά καλά. Το ίδιο ε, στην ε, κεντρική κυβέρνηση. Έχουμε μια ανθούσα τουριστική βιομηχανία. Η οποία πήγαινε τόσο καλά που προσφέρει υψηλά εισοδήματα σε αυτό το τομέα. Όπως ξέρετε έχουμε και διάφορους τομείς στο κυνήγι, ε, διάφορα μέρη όπως το Κιλιμάντζαρο που είναι πολύ σημαντικό όρος, ε, το οποίο επισκέπτονται πολλοί τουρίστες και στην πλευρά της Ανζιβάρης ε, έχουμε πανέμορφες παραλίες με λευκή άμμο όπου είστε όλοι ευπρόσδεκτοι και όπου μπορείτε να απολαύσετε τις λευκές παραλίες. Ο τουρισμός λοιπόν είναι ένα από τους σημαντικότερους, ε, πηγέ τις σημαντικότερες πηγές εισοδήματο για τη Ζανζιβάρη. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αναγκόμες, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει βέβαια η συνεργασία σας με την Κίνα και η Κίνα είχε επενδύσει πέρα από τις ε, παραδοσιακές με ε, μορφές επενδύσεων σε σιδεοδρόμους. Νομίζω ότι έχει κάνει επενδύσεις και σε λιμάνια. Και όλα αυτά έχουν σχέση με την ανακάλυψη φυσικού αερίου. Πώς ε, αξιολογείται αυτή η συνεργασία σας με την Κίνα Πιστεύω και άλλες χώρες αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα. Πώς αντιμετωπίζετε το πρόβλημα της διαφθοράς στη χώρα σας, στην δική σας περίπτωση. Ξέρω ότι έχει επιφορτιστεί τώρα, μάλλον ότι ένας υπουργός έχει χάσει τη θέση του λόγω της διαφθοράς. Και υπάρχει και το πρόβλημα της απαγής γης που συνδέεται με την παραγωγή βιοκαυσίμων που οδήγησε στην παρέτηση αυτού του Υπουργού. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λοιπόν ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση που είχε να κάνει με βιοκαύσιμο και αρπαγηγής. Σας ευχαριστώ πολύ. Η Ταζανία έχει πολλούς φίλους. Μέσα στην Αφρική και έξω και από την Αφρική, στην Ασία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες του κόσμου. Η Κίνα έχει μια μακρά φιλία με την ε, Τανζανία και έχουμε συνεργαστεί μαζί τους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τις περισσότερες φορές έχουμε μια υποστήριξη από την Κίνα που δεν συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Είναι πολύ καλό λοιπόν για μια φτωχή χώρα να μπορεί να πάρει χωρίς όρους οικονομική υποστήριξη όπως αυτή που παίρνουμε από την Κίνα. Αναφερθήκατε στο θέμα της αρπαγής γης στην Τανζανία, σε κάποια τμήματα της ε, Αρούσα συμβαίνει αυτό. Και αγαπητοί συνάδελφοι, το θέμα αυτό αφορά ουσιαστικά την ε, ε, απαλωτρίωση γεών από την κυβέρνηση χωρίς την πρέπουσα αποζημίωση. Το έχουμε αντιμετωπίσει όμως αυτό το θέμα στο νέο σύνταγμα το οποίο θα τεθεί σε δημοψήφισμα κάποια στιγμή τον Ιούλιο του έτους αυτού. Και έχουμε ε, κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να ε, προασπιστούν τα δικαιώματα των ε, γεωργών, των κτηνοτρόφων, των αλλιέων, όλων αυτών που χρειάζονται να έχουν μια σχέση με τη γη και να χρησιμοποιούν την γη και τους υδάτινους πόρους. Όταν λοιπόν η κυβέρνηση χρειάζεται να απαλωτριώσει μια έκταση η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται πραγματικά από βοσκούς ή από γεωργούς το Σύνταγμά μας προβλέπει να δοθεί η αντίστοιχη αποζημίωση, μια επαρκής αποζημίωση, ώστε τα άτομα αυτά να μην αντιμετωπίσουν πρόβλημα με το να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους σε κάποιο άλλο σημείο της χώρας. Ένα άλλο θέμα όμως, το οποίο θέλω να τονίσω είναι το εξή. Αν μια έκταση απαιτείται για να κάνει κάποιο αναπτυξιακό έργο η κυβέρνηση, τότε μπορεί να αντικατασταθεί η γη η οποία απαλατριώνεται με κάποιο άλλο κομματίες, με κάποια άλλη ε, έκταση γης για να αποσημειωθεί ο γεωργός, η τα κτλ. Εάν ναι, αυτό δεν είναι αυτό πρέπει να δοθεί οικονομική αποζημίωση. Και όλα αυτά περιλαμβάνονται στο νέο σύνταγμα το οποίο κάποια στιγμή προς το τέλος Ιουλίου θα τεθεί σε δημοψήφισμα. Πρόεδρε, η αποστολή μου, η αντιπροσωπεία μου, τους βλέπω, Θέλω και αυτοί να πούνε κάτι. Θα μπορούσα λοιπόν με την αδειά σας βέβαια να τους δώσω το λόγο. Ίσως για τα διάφορα ε, θέματα να προσθέσουν κάτι αν έχουν σε αυτά που είπα εγώ. Ο κύριος Ζεώρα ήταν ε, πρωθυπουργός και ήταν και στο σώμα στην ε, Τανζανία. Παρακαλώ. Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε αυτό που ρώτησε ο κ. Τσάρλς Τάνοκ για τον ρόλο της Τανζανίας προκειμένου να διατηρήσει την ειρήνη στην Ανατολική Αφρική. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η Τανζανία για πολλά χρόνια είχε κεντρικό ρόλο στην πολιτική αρένα και στη διπλωματία. Η Τανζανία λοιπόν ενδιαφέρεται πάρα πολύ για την ειρήνη και τη σταθερότητα στις χώρες της περιοχής, στην Ανατολική Αφρική. Για παράδειγμα τον Μπουρούντι. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο πρόεδρος Κουρούνζιζα θέλει να έχει τρίτη θητεία. Κάτι το οποίο οδήγησε σε τεράστιες διαμαρτυρίες στο Μπουρούντι και στην Πουζουμπούρα. Το θέμα όμως είναι... Κοιτάξτε τι λέει η ειρνευτική Συμφωνία της Αρούσα. Λέει σαφώς ότι ο πρόεδρος πρέπει να έχει δύο θητείες. Το πρόβλημα όμως είναι θέμα ερμηνείας. Πώς υπολογίζουμε τις δύο θητείες. Συμφωνήθηκε στην Ειρηνευτική Συμφωνία πέντε χρόνια μεταβατική περίοδος και μετά άλλα πέντε χρόνια μετά τη μεταβατική περίοδο. Γι' αυτό, Κουρούτζη, αυτό που λέει το επιχείρημα του είναι το κατά πόσο η μεταβατική περίοδος αυτή η πρώτη των πέντε ετών συμπεριλαμβάνεται ή όχι στις δύο θητείες. Αυτό είναι το ζήτημα. Κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το θέμα της περιφερειακής εξουσίας. Εμείς δεν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά το θέμα είναι το κατά πόσο η μεταβατική περίοδος υπολογίζεται ή δεν υπολογίζεται. Αυτό είναι το ζήτημα. Εγώ πιστεύω ότι είναι και δικιά μας ευθύνη να καθίσουμε με την κυβέρνηση του Μπουρούντι να εξηγήσουμε το μέγεθος του προβλήματος. Γιατί όσον αφορά την πολιτική σταθερότητα στην περιοχή είναι σημαντικό και η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Πιστεύω ότι θα θέσει σε κίνδυνο όλα τα επιτεύγματα που έχουμε πετύχει μέχρι τώρα. Έρχομαι τώρα στο θέμα της Κίνας. Γιατί η Τανζανία έχει σχέσεις με την Κίνα, τόσο πολλές όσον αφορά την αναπτυξιακή βοήθεια. Η Τανζανία και η Κίνα ήταν πάντα φίλες χώρες. Οι δεσμοί εντάθηκαν τα τελευταία 50 χρόνια. Η Κίνα δίνει αρρωγή στην Ταζανία τη δεκαετία του 60 για παράδειγμα θα θυμόσασταν. Η Κίνα μας έδωσε πάρα πολλά χρήματα για να χτίσουμε τους σιδηροδρόμους και να συνδεθεί η Τανζανία με τη Ζάμπια. Ο δεύτερος λόγος όμως γιατί η Τανζανία έχει αυτές τις φιλικές σχέσεις με την Κίνα είναι ότι η Κίνα τις περισσότερες φορές όταν ασχολείται με τις αφρικανικές χώρες οποιαδήποτε ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο υπόλοιπο κόσμος συνδέει την αναπτυξιακή βοήθεια με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή με θέματα διακυβέρνησης, η Κίνα δεν το κάνει. Προσφέρει αναπτυξιακή βοήθεια στις αφρικανικές χώρες χωρίς να τη συνδέει με θέματα διακυβέρνησης ή με θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οπότε οι αφρικανικές χώρες, οι φτωχές χώρες πιστεύουν ότι αποτελεί καταφύγιο για αυτές προκειμένου να πετύχουν αναπτυξιακή ε, βοήθεια και να κερδίσουν σε ανάπτυξη. Αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι αφρικανικές χώρες έχουν συσφίξει τους δεσμούς με την Κίνα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να απευθύνουν ερωτήσει. Αν όχι, εξοχότατε να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ και ελπίζω ότι όλα όσα είπατε ότι αναμένονται να γίνουν στη χώρα σε πολιτικά θέματα θα γίνουν υπό καλές συνθήκες. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. To be here with you and share with you. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου επιτρέψετε να βρίσκομαι εδώ και να μοιραστώ μαζί σας όλα τα θέματα που συζητήσαμε. Σας ευχαριστώ αξιότιμα μέλη. Ας περάσουμε απευθείας στο επόμενο σημείο. Τη συζήτηση ε, του εγγράφου της ε, κυρίας Γκόμες, ο αντίκτυπος που έχουν εξελίξει οι ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές, τις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη. Η κυρία Γκόμες ζήτησε τη συζήτηση αυτή της εκθεσής της, διότι ουσιαστικά δεν είχαμε την ευκαιρία να γίνει αυτή η συζήτηση στην ΣΕΝΤΕΡ. Θα συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση μέχρι τις 5.30 όπου μετά θα ακολουθήσουν οι ψηφοφορίες και για αυτή την έκθεση αν δεν κάνω λάθος. Κυρία Γκόμες, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία να ακούσω και απόψε ενδεχομένω συναδέλφων που υπάρχουν ακόμα για την έκθεση, αλλά στην παρουσιαφάση θα ήθελα ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους και για την εξαιρετική του συνεργασία. Καταφέραμε να καταλήξουμε σε μεγάλο αριθμό συμβιβασμών επί ουσιοδών στοιχείων. Η συμβολή τους υπήρξε σημαντική και οδήγησε σε τεράστια βελτίωση του δικού μου κειμένου. Θα ήθελα επίσης να επισημάνω, επειδή Συχνά έχουμε τόσους συγκρούσεις αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιτροπών και αυτό αποτελεί τρανό παράδειγμα πρέπει να πω ότι η συνεργασία με την ΕΜΚΟ λειτουργήσε εξαιρετικά. Διότι φυσικά το θέμα αυτό, αντίκτυπος που έχουν εξελίξει στις ευρωπαϊκές αμυντικές αγορές, ε, στις δυνατότητες ασφάλειας και άμυνας στην Ευρώπη, είναι ένα θέμα που εγώ είδα από τη δική μας οπτική γωνία από την ε, οπτική γωνία της υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ δεδομένης και της συζήτηση που θα γίνει μεταξύ των Υπουργών Άμυνα τον Ιούνιο με την προκαταρκτική αξιολόγηση δηλαδή για το πώς οι οδηγίες ε, περί δημοσίων συμβάσεων ε, άμυνας θα υλοποιηθούν. Αλλά φυσικά η πραγματική αξιολόγηση ε, της ε, εφαρμογής θα γίνει του συναδέλφους ε, στην ΙΜΚΟ. Εμείς κάνουμε περισσότερο πολιτική αξιολόγηση και πώς επηρεάζονται οι δυνατότητες ασφαλείας και αμυνάς μας σε εποχές που αντιλαμβανόμαστε πόσο πολύ τις χρειαζόμαστε. Και πρέπει να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο συνεργάστηκα με τον συνάδελφο εισηγητή από την ΙΜΚΟ με τη συνάδελφο εισηγήτρια ήταν εξαιρετική κυρία Κάμπιας κατάλαβε πολύ καλά ότι δεν προσπαθούμε να ποδοπατήσουμε ο ένας αρμοδιότητας του άλλου. Ήταν εξαιρετική συνεργασία γιατί κατάλαβαν από πολλές από τις ανησυχίες μας όπως για το ζήτημα των offset, των, αντισταθμίσεων. Είναι δύσκολο ερώτημα διότι υπάρχουν διάφορες απόψεις ε, όταν ο, οργανισμο, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας ε, παραδέχεται ότι ένας μεταβατικός μηχανισμός εφόσον εστιαστεί ε, στην ισχύση της βιομηχανικής βάσης και της, και της ε, βάσης της τεχνολογικής έρευνας για την Ευρωπαϊκή Άμυνα ενώ η Επιτροπή είχε μια προσέγγιση πιο εστιασμένη και αρνητική για την εσωτερική αγορά. Αλλά οι συνάδελφοι της ΕΜΚΟ αντάλλαξαν απόψεις μαζί μας, χάλι στην εισηγήτρια της ΣΥΜΚΟ και κατάλαβαν πολύ καλά τις δικές μας θέσεις. Έτσι καταφέραμε να καταλήξουμε σε παρόμοια γλώσσα τόσο στη δική μας έκθεση όσο και στην έκθεση της ΣΥΜΚΟ. Γεγονός που θεωρώ σημαντικό διότι θα καταστήσει σαφές το μήνυμα του Κοινοβουλίου. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, ε, το Συμβούλιο και πιστεύω ότι εδώ έχουμε ένα μήνυμα που είναι κατανοητό και σαφές. Εφόσον εγκριθεί από την Επιτροπή μας και μετά από το Κοινοβούλιο, το μήνυμα αυτό θα φτάσει και δεν θα περάσει απαρατηρήτω από τι κυβερνήσεις μας γιατί παρατηρούμε ότι πολλέ κυβερνήσει, όχι όλες, λόγω της οικονομικής κρίσης ε, προβαίνουν σε τεράστιε περικοπές ε, στην άμυνα με σημαντικές συνέπειες. Ακόμα και με υπονομώσεις στρατηγικών τεχνολογιών και επιχειρήσεων στον τομέα, γεγονός που μας ε, θέτει σε κίνδυνο, ενώ άλλες χώρες με καλύτερες οικονομίες ε, ίσως να μην κάνουν τόσες περικοπές αλλά δεν αξιοποιούν ε, ικανοποιητικά τα χρήματα των φορολογουμένων τους διότι ξέρουμε ότι οι δυνατότητες αυτών των αγορών άμυνας ε, προσφέρει πολλές δυνατότητες διαφθοράς κτλ. Χαίρομαι λοιπόν για τη συμβολή όλων και για του συμβιβασμού ε, στου οποίου καταλήξαμε. Πιστεύω θέλουμε ένα σαφέ μήνυμα και το μόνο που έχω να πω είναι ότι ελπίζω το Συμβούλιο να ε, ε, εισακούσει και να δράσει επιτέλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Λέζιν, παρακαλώ. <clears throat> vielen Dank. Ευχαριστώ και εγώ. Ήδη στην πρώτη ανταλλαγή απόψεων που είχαμε κάνει, όπως αναφέρθηκε από την ομάδα μας, την GUNGL, είχαμε εκφράσει τις σοβαρές αντιρρήσεις μας σε σχέση με τα μέτρα και τους στόχους που αναφέρει η έκθεση της κυρίας Αυτό το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα είναι η ενίσχυση της εξοπλιστικής βιομηχανίας, όπως το ανέφερε, και οι προσπάθειες να υπάρξει περαιτέρω ε, βοήθεια της έρευνας για τα εξοπλιστικά με υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είναι ένα θέμα που <clears throat> έχει τεθεί και από την Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει προγράμματα επιδοτήσεως στην εξοπλιστική βιομηχανία, κάτι το οποίο η πολιτική μου ομάδα το απορρίπτει διαρρήδη. Υπάρχουν κάποια άλλα σημεία, το σημείο 12 και 13 που πρέπει να τα απορρίψω, ε, συγγνώμη, πρέπει να τα να συμφωνήσω μαζί τους ό,τι αφορά την ε, κριτική για την έλλειψη ελέγχου των εξαγωγών εξοπλιστικών συστημάτων. Αλλά και στο σημείο αυτό εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ περισσότερο στα σημεία αυτά για τα σημεία 12 και 13 που αφορούν τους ελέγχους εξαγωγών εξοπλιστικών συστημάτων. Έχουμε λοιπόν αρκετά διαφορετική γνώμη, αλλά σας λέω και πάλι, γενικά η κατεύθυνση αυτής της έκθεσης είναι κάτι το οποίο το απορρίπτει η ομάδα μας, δεν υποστηρίζει την ε, δημιουργία περισσότερων εξοπλιστικών συστημάτων. Εμείς αντίθετα θέλουμε να υπάρξει αφοπλισμό σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωση. Γιατί πρέπει να τονίσουμε ότι όλα αυτά επηρεάζουν και τα δημοκρατικά καθεστώτα. Υπάρχει μείωση του δημοκρατικού ελέγχου λόγω της πίεσης του εξοπλιστικού τομέα, ο οποίος αυξάνει την επιρροή του. Το αποτέλεσμα είναι ότι ότι κινδυνεύει η δημοκρατία σε πολλές χώρες εάν δεν υπάρξει μία μείωση των εξαγωγών εξοπλιστικών συστημάτων. Και έχουμε γι' αυτό το λόγο εκφράσει τις θέσεις μας και το έχουμε αναφέρει και στην γραμματεία. Ο κύριος Μπουτικόφερ. Πάρα πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Πρώτα απ' όλα, Θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Γκόμες για την ποιότητα της συνεργασίας μαζί μας. Νομίζω ακόμα και οι συμβαστικές τροπολογίες που επετέφθησαν είναι θετικές. Τρεις παρατηρήσεις μονάχα θέλω να κάνω που συνδέονται και με αυτά τα οποία είπε η κυρία Λέζινγκ προηγουμένως. Όπως και στο παρελθόν λοιπόν εμείς ως πράσινοι πιστεύουμε ότι δεν πρέπει να χρηματοδοτηθεί η αμυντική έρευνα από τον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, για μένα αυτή η έκθεση είναι μια ευκαιρία να προχωρήσουμε σε μια μείωση των ε, εξαγωγών οπλικών συστημάτων, ένας από τους λόγους για τους οποίους δεν μπορώ να υποστηρίξω αυτήν την έκθεση. Και τρίτον, δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια μορφή συσχετισμού μεταξύ του ύψους των εξοπλιστικών δαπανών και της στρατιωτικής ικανότητας. Άμα δω πόσα είναι τα εξοπλιστικά προγράμματα στη Γερμανία τα τελευταία χρόνια που καταδαπάνησαν απίστευτες ε, πιστώσεις αλλά δεν έχουν δημιουργήσει αμυντική ικανότητα. Πρόκειται για μια κατασπατάληση χρημάτων. Δεν υπάρχει άλλο τομέα στην Ευρώπη όπου να έχουν καταδαπανηθεί και κατασπαταληθεί τόσα χρήματα όσο ο αμυντικός τομέας. Εγώ νομίζω ότι με πολύ λιγότερα χρήματα θα μπορούσαμε να έχουμε πιο απο, αποτελεσματικές αμυντικές ικανότητες και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Γκάλερ, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ, λέει ο κ. Γκάλερ. Συγγνώμη που καθυστέρησα να έρθω. Θέλω να εκπροσωπήσω και τον συνάδελφο κύριο Κίρτσο, ο οποίος είναι ο σκηριώδης εισηγητής για το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω και προσωπικά και εξορμαστού κυρίου Κίρτσου την κυρία Γκόμες για την πολύ καλή συνεργασία και για το <clears throat> αποτέλεσμα που έχει επιτευχθεί με τις 14 τροπολογίες συμβιβασμού. Για μένα είναι μια πολύ καλή και εξισορροπημένη έκθεση. Έχουμε διαπιστώσει όλοι μαζί ότι μέσα στην ε, χρηματοπιστωτική κρίση που περνάμε, την οικονομική κρίση, υπάρχουν περικοπές οι οποίε οδήγησαν σε μια μείωση της αμυντικής ικανότητα των χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και δεν έχουμε βρει τις απαραίτητες ε, απαντήσεις ως Ευρωπαϊκή Ένωση για πάρα πολλέ προκλήσεις και απειλές στον περίγυρό μας. Έχουμε τονίσει την ανάγκη να έχει στρατηγική αυτονομία η Ευρωπαϊκή Ένωση και να εξασφαλίσει την ασφάλεια εφοδιασμού και επειδή πολλές φορές τίθεται ένα ερωτηματικό εικόνα το κεφάλι τους με απορία ορισμένα όταν μιλάμε για στρατηγική αυτονομία αναφέρομαι στις αποστολές για τις οποίες έχουμε συμφωνήσει και όλοι μας. Δηλαδή όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτελεί τέτοιες αποστολές θα πρέπει να έχει αυτονομία. Δεν μιλάμε για αυτονομία έναντι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Δεν πρέπει να κάνουμε αποστολές εναντίον του ΝΑΤΟ ή των ε, Πολιτειών. Αλλά όταν εμείς αποφασίζουμε ομόφωνα να εκτελέσουμε κάποιες αποστολές θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα ε, να τις υλοποιήσουμε με τα δικά μας μέσα. Αυτή είναι η στρατηγική αυτονομία. Εξακολουθεί λοιπόν αυτό να παραμένει μια πρόκληση για μας και απαιτεί την περαιτέρω εξέλιξη της βιομηχανικής μας βάσης στον τομέα των εξοπλισμών. Ελπίζουμε λοιπόν ότι η συνολική δέσμη μέτρων για τα αμυντικά θέματα θα μπορέσει να προωθήσει και μεγαλύτερη συνεργασία στον τομέα αυτό των εξοπλισμών στην Ευρώπη. Πιστεύω περαιτέρω ότι με την έκθεση αυτή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς στην καλύτερη προετοιμασία της ε, διάσκεψης κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων τον Ιούνιο του 2015. Με τον τρόπο αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχει ζητήσει να υπάρξει μια διάσκεψη κορφής και για τα αμυντικά θέματα. Μπορούμε να έχουμε μια ελπίδα ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα υλοποιήσουν αυτή τη στρατηγική και έτσι θα βρίσκεται καλύτερα εξοπλισμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αντιμετωπίσει υποκλήσεις και απειλές. Επίσης, έχουμε μια θετική αντιμετώπιση για το έργο του Ευρωπαϊκού Φορέα Άμυνας, ΕΝΤΑ, και της ε, δράση τη Κομισιόν για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού. Ελπίζουμε λοιπόν ότι και αυτό θα είναι ένα προεξάρχον θέμα κατά την διάσκεψη κορυφής του Ιουνίου και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε περισσότερο από ότι επετέχθη στο προηγούμενο Συμβούλιο που αντιμετώπισε τα θέματα άμυνας. Ελπίζουμε ότι τον Ιούνιο θα μπορούμε να <clears throat> εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια εφοδιασμού για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω λοιπόν θα υπάρξει μια βρήκα πλειοψηφία που θα υποστηρίξει το έργο της εισηγήτριας. κύριος Ευχαριστώ πολύ. Είναι θετική έκθεση που υπογραμμίζει ότι χρειάζεται μια αυτονομία τεχνολογίας μεταξύ άλλων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όμως, θα έπρεπε να υπάρχει και μια ευρωπαϊκή άμυνα. Για να υπάρχει όμως μια ευρωπαϊκή άμυνα θα πρέπει να έχουμε και μια κοινή άποψη και θα πρέπει να συμφωνούμε μεταξύ μας για τις πρόπτικες και για το τι πρέπει να προστατεύσουμε. Η ευρωπαϊκή άμυνα όμως δεν υπάρχει. Το διαπιστώνουμε κατά τη διάρκεια των σημερινών κρίσεων. Δεν υπάρχει κοινή άποψη, κοινή προσέγγιση, ιδιαίτερα μεταξύ των μεγάλων χωρών. Έπειτα, η έκθεση αυτή εισφάλει και εδώ θα μιλήσω σαν ειδικό γιατί, γιατί υποθέτει έκθεση ότι αν βάλουμε από κοινού τους πόρους μας θα μας κοστίσει λιγότερο. Μα όχι. Το φάλει για παράδειγμα σε σχέση με το Eurofighter ή σε σχέση με το GFS. Επειδή δεν βάλαμε μαζί τους πόρους μας γι' αυτό η Γαλλία έκανε ένα καλό αεροπλάνο. Αν είχαμε κάνει το αντίθετο θα μας είχε κοστίσει πολύ περισσότερο. Η σχέση ανάμεσα στο Eurofighter και το Rafale είναι 1 προς 5. Και δεν μιλάω για το GSF ή το ESF-15 γιατί εκεί είναι 1 προς 40. Δεν είναι επειδή θα έχουμε κοινή άμενα που θα μας στοιχήσει πιο φτηνά. Αυτό δείχνει η εμπειρία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Γκόμες. Αν δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο. Παρακαλώ κυρία Γκόμε. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές για τα σχόλιά τους, τα ουσιαστικά ο σχόλιά τους. Την κυρία Λουζίν, θέλω να πω, δεν μου κάνει εντύπωση που η ομάδα της έχει αναλλακτική έκθεση, μπορεί όμως να συμφωνήσουμε με μερικά από αυτά που ανέφερε. Γιατί βέβαια η βασική διαφωνία μας είναι ότι δεν πιστεύει ότι χρειάζεται μια ευρωπαϊκή άμυνα, ενώ εγώ, η ομάδα μου, όπως και άλλοι, πιστεύουμε ότι χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή άμυνα. Και πιστεύουμε επίσης ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να βάλουμε τις δυνάμεις μας από κοινού και να αποκτήσουμε τη στρατηγική αυτονομία όχι με αρνητικό τρόπο, αλλά με έναν τρόπο που να μας επιτρέπει να δράσουμε εφόσον κρίνουμε ότι πρέπει να δράσουμε, βάσει βέβαια των αξιών και αρχών μας. Εγώ πιστεύω σε μια ευρωπαϊκή άμυνα η οποία στηρίζεται στις αρχές και στις αξίες μας. Και γι' αυτό και υποστηρίζω μια αποστολή SPC στην Μεσόγειο για να σωθούν ζωές ή όπως κάναμε για να αντιμετωπίσουμε την πειρατεία στον ειδικό, γιατί να μην κινητοποιήσουμε τα δικά μας σκάφη και την ακτοφυλακή και τις ενεργείς δυνάμεις μας για να σώσουμε ζωές ε, που γίνονται ανθρώπων που είναι θύματα εκείνων των διακινητών. Εντάξει κυρία Αλέζιν και εγώ δεν συμφωνούμε, μάλλον όσον αφορά τα μέσα. Επίσης θέλουμε να πιάνουν τόπο τα λεφτά μας και θέλουμε διαφάνεια. Θέλουμε να ξέρουμε πού πάνε τα χρήματα. Εγώ, για παράδειγμα, δεν πιστεύω ότι τα χρήματα που δίνουν για τα πυρηνικά κάποιες χώρες εξυπηρετούν. Γιατί δεν πιστεύω ότι τα πυρηνικά είναι αποτρεπτική δύναμη. Αντίθετα, εγώ θα ήθελα να δίνουμε τα χρήματά μας αλλού εκεί που πιστεύω εγώ ότι έχουμε ανάγκη. Αλλά εντάξει, υπάρχουν διαφωνίες, το καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πάντω για τα σχόλια την κυρία Τώρα, κύριε Μπουτικόφερ, χαίρομαι που αυτή τη φορά συμφωνούμε και σα ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια στοιχεία, κάποια θεμελιώδη, αλλά σίγουρα θέλουμε να πιάνουν περισσότερο τόπο τα χρήματά μας. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε, ότι δεν υπάρχει σχέση ανάμεσα στα χρήματα που δίνουμε και τη στρατιωτική ικανότητα που έχει κάθε χώρα. Συμφωνώ μαζί σας. Και ακριβώς γι' αυτό είναι που λέω ότι χρειαζόμαστε μια κοινή ευρωπαϊκή λογική για το θέμα αυτό γιατί έτσι θα καταλάβουμε καλύτερα ποιες είναι οι ικανότητες που χρειαζόμαστε, όχι μόνο τώρα αλλά και στο μέλλον και θα συνεργαστούμε για να αποκτήσουμε τις ικανότητες αυτές που μερικές φορές δεν αντιστοιχούν σε αυτές που αναπτύσσουν οι κυβερνήσεις μας μερικές φορές στενόμυαλα. Το καταλαβαίνουμε. Η κυβερνοασφάλεια, για παράδειγμα, είναι πολύ βασικό στοιχείο, όχι μόνο για την εσωτερική ασφάλεια, αλλά και για την άμυνα και αντιλαμβανόμαστε ότι δεν έχουμε ακόμα τα μέσα για αυτή την κυβερνοασφάλεια. Γι' αυτό νομίζω ότι έχει νόημα να δουλέψουμε με ευρωπαϊκή προσέγγιση από κοινού και τα άλλα, offsets κλπ. Όντω χρειαζόμαστε περισσότερα. Κύριε Γκάλερ, ευχαριστώ πολύ για αυτά που είπατε. Και πάλι μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια σημεία, αλλά συμφωνούμε σε πολλά θεμελιώδη. Και νομίζω ότι η αντίληψή μας, ο τρόπος που καταλαβαίνουμε εμείς τη βιομηχανική βάση για την άμυνα στην Ευρώπη είναι ίδια. Αν δεν το κάνουμε ευρωπαϊκά δεν θα το κάνουμε καθόλου. Και χρειαζόμαστε έρευνα και ανάπτυξη και στην κυβερνοσφάλεια αλλά και αλλού. Πιστεύω λοιπόν πραγματικά, κοιτάξτε όλοι το γνωρίζουμε, πριν από λίγα χρόνια καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι εξαρτιόμαστε από τα ρωσικά Αντόνοφ για να μπορούμε να κάνουμε αποστολές ε, CFCP. Τώρα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα από ό,τι ήταν τότε. Εδώ χρειαζόμαστε αυτονομία. Τέλος, κύριε Σαφάζολαν, χαίρομαι που δεν συμφωνείτε, που επικρίνετε την έκθεσή μου. Αλλιώς θα ανησυχούσα αν συμφωνούσατε συνέπειπτα οι απόψεις σας με τις δικές μου. Δεν συμφωνώ με τη δικιά σας λοιπόν την άποψη. Μπορεί Πράγματι, κάτω από ορισμένε συνθήκες, κοινά προγράμματα να κοστίζουν περισσότερα. Αλλά αυτό, αν έγινε, έγινε γιατί δεν έγιναν σωστά τα πράγματα. Διότι αν έχουμε κοινά προγράμματα, αν μη τι άλλο, χρησιμοποιούμε την ε, βασική βιομηχανική δομή. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να βοηθήσουν. κυβερνοχώρος και αλλού οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Αλλά εξαρτάται πώς γίνεται η διαχείριση. Δεν αρκεί να έχουμε ένα κοινό σχέδιο, πρέπει να ελέγξουμε το κόστος. Και γι' αυτό ακριβώς είναι που χρειάζεται ένας χώρος ευρωπαϊκός άμυνας. Ας ψηφίσουμε. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα συναδελφοί έχουμε τρεις εκθέσεις ε, που θα ψηφίσουμε και ξεκινάμε με την έκθεση που μόλις συζητήσαμε, την έκθεση της Ανά Γκόμες. Ετοιμαστείτε λοιπόν, ε, βάλτε τις κάρτες στις υποδοχές και αν συμφωνείτε όλοι και είστε έτοιμοι και ο κύριος Πρέντα. Ωραία. Λοιπόν, περνάμε στην ψηφοφορία έκθεση της Ανασγκομές. Έχουμε τη συμβιβαστική 1, ποιος είναι υπέρ, κατά, ε, αποχές, εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 49. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πριν από τροπολογία 63 υπέρ, 62 συγγνώμη, Κατά τμήματα ψηφοφορία, πρώτο τμήμα της 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Δεύτερο τμήμα λοιπόν της τροπολογίας 62, άρχεται η ψηφοφορία. Περιμένουμε. okay. Είναι εντάξει. Ωραία, πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παίρναμε στην τροπολογία 63 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στην 72. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 73 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές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 αποχές ας το ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την τροπολογία 106 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορία. ψηφοφορίας εγκρίνεται συν μία κάποιος που δεν ψήφισε ηλεκτρονικά περνάμε στην 107 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 κατά τμήματα ψηφοφορία, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα υπέρ, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την 124 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 125-126 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 ε, υπέρ κατά καταπίπτει καταπίπτει επειδή 125 και 126 απορρίφθηκαν ε, εγκρίθηκαν συγγνώμη 128 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά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 και περνάμε στην τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. One more. Άλλη μια ψήφος, πέρας ψηφοφορίας. Συγχαρητήρια, κυρία Γκόμες. Η κυρία Λέζινγκ θέλει να σας πει κάτι. Έχετε το λόγο. Ναι. Το ανέφερα ήδη, αλλά απλώς ήθελα να πω ότι καταθέτουμε μια έκθεση μειοψηφία. Ευχαριστώ πολύ, ο Πρόεδρος. Περνάμε στις επόμενες εκθέσεις. Για την ε, Μαύρη Θάλασσα. Τη στρατηγική κατάσταση στη Μαύρη Θάλασσα. Είσαστε όλοι έτοιμοι. Λοιπόν, έκθεση για την ε, Μαύρη Θάλασσα. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνητες. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 109 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 σε τέσσερα τμήματα τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές δεκτό δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές πρέπει να ελέγξουμε για το δεύτερο τμήμα της 111 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπάρχει ένας πλεονάζων στους μη εγγεγραμμένους. πρέπει ένα από του μη εγγεγραμμένου να μην ψηφίσει. Βγάλτε μία κάρτα. Ρίξτε το κοροναγράμματα αν θέλετε. Δεν μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα όσο δεν ε, ψηφίζεται όσο, όσο είναι κάποιος παραπάνω που ψηφίζει. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σιάφρα. Απορρίπτεται λοιπόν. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται τέταρτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές ελέγχουμε. Τέταρτο τμήμα. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Και πάλι ένας παραπάνω από τους μη εγγεγραμμένους. Πέρα της ψηφοφορίας απορρίπτεται. <coughs> όχι, όχι, συγγνώμη. Περνάμε στην 112. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 118. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 115 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 114 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 121 και 122 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 124 υπέρ κατά αποχές. Ελέγχουμε την 124. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 125. Υπέρ. 125 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 137 <clears throat> υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 149 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 152 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Προφορική τροποποίηση του εισηγητή που αναφέρεται στο τέλος καταλόγου. Η 152 δεν έχει εγκριθεί, οπότε μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία του εισηγητή. Κατά αποχές για την προφορική τροποποίηση, μάλιστα. Ας ελέγξουμε λοιπόν για την προφορική. 152 λέει ο πρόεδρος, συγγνώμη, προφορική τροποποίηση, προφορική τροποποίηση. Άρχεται η ψηφοφορία. Είναι στο τέλος του καταλόγου ψηφοφορίας. Αν επιμένετε μπορώ να σας τη διαβάσω κιόλας. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι πρωτοβουλίες συνεργασίας για την περιφερειακή ασφάλεια της Μαύρης Θάλασσας, Black Sea 4 και Black Sea Harmony, που έχουν σαν στόχο να δείξουν προς τον έξω κόσμο ότι οι παράκτιες χώρες μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους και η προσθήκη είναι εδώ. Ενώ διατηρούν την ικανότητά τους για να αναζωογονήσουν την μελλοντική συνεργασία μεταξύ των χωρών αυτών, είναι τώρα όμως σε κατάσταση παράλυσης. Δηλαδή η Black Sea και η Black Sea Harmony. Εντάξει. Άρχεται η ψηφοφορία. για την προφορική τροπολογία 1. Ψηφίστε όπως θέλετε. Πέρας. Μια στιγμή. Εντάξει. Εγκρίνεται. Σύμβασκη 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Σύμβασκη 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ...179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται... ...181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 191 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 192 όχι δεν, δεν, χρειάζεται να ψηφίσουμε εκπίπτει το ίδιο και 193 196 υπέρ κατά αποχές έλεγχος για την 196 άρχεται η ψηφοφορία Πάλι περισσεύει ένας από τους μη γεγραμμένους. Ε, εντάξει. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Πέρας. Απορρίπτεται. 197 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 198 εκπίπτει. Συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 209 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 210 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η 211 εκπίπτει, η 212 επίσης. 214. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δύο υπέρ κατά αποχές γκρίνεται, δύο δεκαέξι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 17 υπέρ συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2, Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 2.26 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 2.28 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 2.29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 2.30 ναι, εκπίπτει, εκπίπτει. Συμβαστική 18 υπέρ κατά Αποχέ. εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. 2.38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.39 και 2.40 οι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 2.44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται απορρίπτονται 2.42 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 2.43 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστή 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 45 υπέρ κατά αποχές συγκρίνετε 2.47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.48 υπέρ κατά απορρίπτεται 2.50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.51 υπέρ κατά αποχές απορρίζεται προφορική τροπολογία 2 ο κύριος Μπουτικόφερ εγώ αντιτίθεμαι στο να ψηφιστεί η προφορική τροπολογία 2 και το εξηγώ κάνει μια δήλωση για, τα, για την πραγματικότητα που δεν έχει καμία σχέση. Το ΝΑΤΟ δεν είχε καμία αεροπορική και ναυτική υπεροχή στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Το να πούμε ότι θα πρέπει να διατηρήσει αυτή την υπεροχή, αυτό δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια ανοησία και φυσικά και εγώ είμαι εναντίον της πολιτικής που εκφράζεται σε αυτή την τροπολογία, την οποία εμείς απορρίπτουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να ψηφιστεί μια τροπολογία που δεν στέκει. Ωραία, δεν την ψηφίσουμε, λέει ο Προχωρούμε. Αν συζητήσουμε τώρα για την ε, υπεροχή του ΝΑΤΟ στην ε, Μαύρη Θάλασσα, μπορεί κάποιο να η να επιχειρηματολογήσει προ την κατεύθυνση αυτή. Δεν σημαίνει ότι επειδή λέει κάποιος από του πράσινου ότι δεν ε, έχουμε υπεροχή. Ευλακίες είναι αυτά, λέει ο κύριος, ο ταξίαρχος Βανόντου. Εάν υπάρξει ανεξάρτητα από το αν συμφωνείτε ή όχι, Υπάρχει διαδικασία για την απόρριψη μια προφορική τροπολογία και αυτό επικαλούμε, λέει ο κ. Μπουτικόφερ. Θα ήθελα να μπω στη συζήτηση, λέει ο πρόεδρος, αλλά δεν μπορώ ως πρόεδρος. Α, τότε ψηφίζουμε το αρχικό κείμενο. Ούτε, ούτε, ε, εντάξει, καλά. Δεν ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρος. Δεν ψηφίζουμε. Χωρίς μικρόφωνο παρέμβαση. Το αρχικό κείμενο παραμένει γιατί η προφορική τροποποίηση δεν μπορεί να ψηφιστεί. Εντάξει. 2.52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε 32 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 36. Κάποιοι κουράζονται, δεν σηκώνουν τα χέρια τους. Πέρας. Απορρίπτεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 42. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτουται, 39 υπέρ κατά αποχές απορρίπτουται, 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτουται, 45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτουται, 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 47 Συγγνώμη, η 44 έχει εκπέσει. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 εξέπεσε. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σύμβαστη 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 60 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική αναφορέ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 3 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οι έξι εκπίπτει, όλες αυτές εκπίπτουν, εννέα, υπέρ, κατά, αποχές, ας ελέγξουμε για την εννέα, άρχεται. Πέρας, απορρίπτεται. Και τώρα πρέπει να γυρίσουμε πίσω γιατί είχαμε πηδήξει την τροπολογία 194. Στην παράγραφο 15 η τροπολογία 194 του κυρίου Τόνι Πικούλα Εντάξει, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Και η τελική ψηφοφορία τώρα. Η ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Εγκρίνεται. Συνεχίζουμε και περνάμε στην τελευταία έκθεση που έχουμε να ψηφίσουμε σήμερα. Γνωμοδότηση είναι, ο συντάκτης γνωμοδότησης είναι ο κύριος Ντανζό. Είσαστε όλοι έτοιμοι να ψηφίσουμε. Τροπολογία 34-35 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Οπότε ψηφίζουμε μαζί το μπλοκ 1. Ποιοι είναι υπέρ της ομάδας Ευρωπαϊκών. Κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία θα ελέγξουμε. Κάποιος κουράστηκε μάλλον και ήθελε κάτι να κάνει. Τώρα το 7 υπέρ, το μπλοκ 7 κατά, αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε, ωραία, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Α, ένας ακόμα. Ωραία. Εγκρίθηκε. Οπότε τώρα πάμε στο μπλοκ 12. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπλοκ 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 86. 86 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 86. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας της οφορίας εγκρίθηκε. 88 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφτεται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 91 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπλοκ 6 υπέρ, κατά, πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το μπλοκ 6. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας ψηφοφορίας Εγκρίθηκε. 93 τώρα υπέρ. Κατά. Κύριε Μποτικόφερ, μπορούμε να συνεχίσουμε παρακαλώ. Πρέπει να συνεχίσουμε. Ο κύριος Μποτικόφερ εκτός μικροφώνου έκανε παραβάση. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 101 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπλοκ 3 υπέρ παρακαλώ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 127 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 129 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Α, να ελέγξουμε, ωραία. Ψηφίζουμε, μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Αν δεν σηκώνετε τα χέρια σας και τα λοιπά, τα ξέρετε. 50... Όχι. 107 ψηφίζουμε τώρα. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. 107. Ξανά, 107 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Εκτός μικροφώνου παρέμβαση, δεν την ακούμε. Ωραία, 59 τότε. Πάμε στην 59. Υπέρ παρακαλώ, 59. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία. 107. Μπορείτε να ψηφίσετε. τη ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 110 τώρα. Υπέρ. Α, λάθος. 108 διορθώνει ο πρόεδρος. 108 Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 113 υπέρ. Α, α όχι, είναι το μπλοκ 13. Μπλοκ 13. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 145 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι σαφές το αποτέλεσμα. 114 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 115 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117-118 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 122 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 123 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 132 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 134-135 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. ηλεκτρονικά ψηφίζουμε 134-135. Ψηφίσατε. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 139 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 140 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 147 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 150 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται απορρίπτεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 153 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 167 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 162 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 162. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα της φοφορίας εγκρίνεται. Τώρα 168. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 169 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπλοκ 4. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Α, θα ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε για το μπλοκ 4. Πέρα στις φοφορίες. Εγκρίθηκε. 163. Υπέρ, κατά, αποχές, θα 163. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις Εγκρίνεται. 164. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Από εδώ το βλέπω καθαρά. Λοιπόν, 165 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 170 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Μπλοκ 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 188. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 176. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 176. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. Μπλοκ 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. 10 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίφθηκε. Να ελέγξουμε. Καλώς. Για το 10, έτσι. Για την ομάδα ψηφοφοριών 10. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρασε ψηφοφορίες. Εγκρίνονται. Εγκρίνονται. Το μπλοκ 10. Εγκρίθηκε. Τώρα καταπίπτουν κάποιες 179 πρέπει να ψηφίσουμε υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 179. 179. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρασε ψηφοφορίες. Απορρίφθηκε. 180 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 83 υπέρ, καταπίπτει. 183 καταπίπτει. Δεν την ψηφίζουμε. 181 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 181. Εκτός μικροφώνου ο κύριος Στάνοκ, δεν τον ακούμε. Δεν ήτανε, λέει ο πρόεδρος, σαφές. Γι' αυτό ζήτησα να ελέγξουμε για την 181. 181 λοιπόν ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Εγκρίθηκε. Θα επιβραδύνω την ψηφοφορία, λέει ο Πρόεδρος, σας υπόσχομαι. Θα πηγαίνω πιο αργά. Συμφωνούμε εδώ τώρα, ναι ή όχι. Ποια σας προκαλεί πρόβλημα. Καλά, μέχρι να τελειώσουν οι διαπραγματεύσει συνεχίζουμε. 182 υπέρ, κατά, αποχές, το ίδιο όπως και άλλη ψηφοφορία. Αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 182. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρες ψηφοφορίε. Εγκρίθηκε. Βλέπετε, η πλειοψηφία είναι υπέρ. 183 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 184 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρα στις ψηφοφορίες, εγκρίθηκε. Υπάρχει πλειοψηφία από ό,τι φαίνεται. 186 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 189 υπέρ, κατά, αποχές. Μ, εδώ πρέπει να ελέγξουμε. 189. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Πέρες προφορίας. Απορρίφθηκε. Τώρα. 190 υπέρ. Υπέρ της 190. Κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Καλώς. Ελέγχουμε για την 190. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας τη φοφορίες, απορρίφθηκε. Με τον άνεμο. 61 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε. 62 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την 62. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλειωσε η ψηφοφορία. Απορρίφθηκε. 191 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 192 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπλοκ 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 195 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε. 196 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε προφορίες, εγκρίθηκε. 197 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 198 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 200 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε για τη 200. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη 200. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε φορείας. Απορρίφθηκε. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 204 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 32. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 208. Υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 208. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 209. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 210 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 211 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 213 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 214 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 214. Ψηφίστε παρακαλώ. Το αποτέλεσμα αλλάζει, δεν είναι πάντα το ίδιο. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίθηκε. 214 ήταν αυτή. «215 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 216 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 218 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Πέρα της ψηφοφορίας. Διαφορά. Τσίμα, τσίμα. Να λέξουμε πάλι θέλετε. Απορρίφθηκε βέβαια. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 220. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 221 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 222 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 223 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 224 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 225 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ, Κατά, δεν είπα το κατά στην 1, λέει ο πρόεδρος. Τώρα, στη 2, κατά. Είμαστε στη 2. Υπέρ παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ της Κατά της 2 εγκρίνεται. 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 39. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. 39. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας τις ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 41. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43. Υπέρ. Κατά θα ελέγξουμε. 43. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 44. Υπέρ. Θέλετε να ελέγξουμε. Κύριε Καστάλντο, άντε για σας εντάξει. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. 42. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Να. Ορίστε. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 47. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 όχι, 48 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ 49. Θέλετε να ελέγξουμε και τη 48. Καλά. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 48. Ψηφίστε. Πέρασε τη ψηφοφορίες. Εγκρίθηκε. Τώρα. 49. Υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 52 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ κατά αποχές θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά, ψηφίζουμε για την 63 παρακαλώ, ψηφίστε. Ψηφίστε. Πέρας της φοφορίας. Απορρίφθηκε. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 72 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 73 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 75-76 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ, κατά, αποχές Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Μπορείτε να ψηφίσετε. Πέρας της σοφορίας, απορρίφθηκε. 78 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται τελευταία ψηφοφορία. 36 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. 36. 36. η τελευταία τροπολογία. Τελευταία, τελευταία. Πέρα τη φοφορίας απορρίφθηκε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τώρα το σύνολο του κειμένου. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρα στις φοφορίες. Συγχαρητήρια, κύριε Τανζό. Κυρίε και κύριοι, αύριο 8 και 30 αρχίζουμε. 8 και 30 αύριο το πρωί. Μακάρι να μπορούσα να το αλλάξω, αλλά δεν γίνεται. 8 και 30 αρχίζουμε αύριο. Καλό βράδυ.